La Επαναλαμβάνονται οι εργασίε. Θα ήθελα να σας μιλήσω για μια διάσκεψη στην οποία χθες συμμετείχα κατόπιν πρόσκλησης ε, του Επιτρόπου Έτιγκερ. Το θέμα ήταν το μέλλον των οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόντες ήταν και άλλοι εξημών και σε διάρκεια ενός πάνελ απάντησα και σε ερωτήσεις της συντονίστριας. Ο Επίτροπος Έτιγκερ επιβεβαίωσε χθε στη διάσκεψη αυτή τα λόγια τα οποία είχε εκφέρει και ενώπιν της Επιτροπής μας. Ότι δηλαδή είναι αποφασισμένος να υπάρξει συμφωνία για ένα πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021, 2026, 2028 την άνοιξη του 2018 το οποίο συνεπάγεται ότι συγγνώμη, την άνοιξη του 2019 λέει ο Άρα το Μάρτιο του 18 θα πρέπει η να έχει καταθέσει την πρότασή της για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ήταν παρόντες ε, τρεις υπουργοί και ένας πρέσβης εκπροσωπούσαν τέσσερις διαφορετικές χώρες μέλη της Ένωσης. Και τα λόγια τους ήταν άκρος ενθαρρυντικά για τους ίδιους πόρους, την ανάγκη επανεξέτασης ε, του προϋπολογισμού. Είπαν ότι θα πρέπει να θεσπιστούν κονδύλια για κατεπήγουσα ε, κατεπίδουσες αποστολές σε θέματα ασφάλειας, μετανάστευσης κτλ. Δηλαδή, η δέσμευση και η προσήλωση στους στόχους ήταν έντονη. Χωρίς να θέλω βέβαια να δεσμεύσω την Επιτροπή μας, είπα ότι το Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να ξεκινήσει μια συζήτηση, αλλά με την προϋπόθεση ότι αμελητή θα συμμετάσχει, θα να συμμετέχει σε όλες αυτές τις συζητήσεις και ιδίω με την προϋπόθεση ότι και οι αρχικοί κρατών και κυβέρνησεων θα μας πούν ποιο είναι το όραμά τους για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα σχέδιο για την Ευρώπη. Και θα πρέπει να κλείσουμε τα διδάγματα και τα συμπεράσματα. Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά, Ίσως μειωθούν οι πόροι που ο Επίτροπος λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν είναι σαφές πότε βέβαια. Κατά πάσα πιθανότητα όμως από το 2019 και μετά η Μεγάλη Βρετανία δεν θα συμμετέχει στον προπολογισμό που σημαίνει ότι θα πρέπει να βρεθούν κονδύλια για να αντισταθμίσουν αυτό το κενό. Μίλησε για περιορισμό σε κάποιες δαπάνες και για μια πρόσθετη συνεισφορά σε νοπό χρήμα από τα κράτη-μέλη. Φυσικά για όλα αυτά τα ζητήματα θα πρέπει άμεσα να ενημερωθούμε για το τι πιστεύει το Συμβούλιο. Θα ήταν χρήσιμο, πιστεύω, σε μια πρώτη φάση να υπάρξει συμφωνία επί του οράματος της Ευρωπαϊκής Φιλοδοξίας, του Ευρωπαϊκού Σχεδίου. Και από εκεί και πέρα να αντλήσουμε και τα δημοσιονομικά συμπεράσματα. Χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία Κάτι που δεν σημαίνει όμως ότι θα υπάρχει αυτό το δημοσιομικό στερέωμα ή γαλαξίας. Δηλαδή τα διάφορα transfer, διάφορες μεταφορές πιστώσεων και άλλα χρηματοδοτικά μέσα που θα καταστήσουν ακατάληπτο τον προπολογισμό της Ένωσης για τον απλό πολίτη. Εμείς νομίζουμε ότι θα πρέπει να μπορούν οι πολίτες να καταλαβαίνουν τι εστί και ευρωπαϊκός προπολογισμό. Εδώ υπάρχει λοιπόν μια δυσκολία πραγματική. Δηλαδή αν δεν υπάρχουν πόροι, πολύ δύσκολα θα μπορέσουμε να καταφύγουμε σε αυτά τα πολλαπλά εργαλεία που καταλήγουν, όπως είπα, σε αυτό το στερέο, σε αυτό το γαλαξία και είναι και κάπως ε, δύσκολο να τα ελέγξουμε ε, κοινοβουλευτικά εμείς. Δεν ξέρω αν ο κύριος Όλμπριχτ, ε, κυρία Γκαρθιά Θάμπαλ, που ήταν επίσης παρόντες και οι δύο σε, αυτό, σε αυτή την διάσκεψη, αν θέλω να μας πούν τις απόψεις τους. Κυρία Γκαρθιά Θάμπαλ, ευχαριστώ εσείς συνοψίσατε πολύ καλά αυτά που ακούσαμε ιδίω το βράδυ. Πράγματι, στο πάνελ που ως πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτών ήσασταν παρόν. Ήταν εφαρυντικά αυτά που ακούσαμε, ήταν και εκπρόσωποι των κυβερνήσεων που είπατε εκεί και έκαναν κάποιες προτάσεις που σε αρκετά μεγάλο βαθμό είναι στην ίδια γραμμή, στο ίδιο μήκο κύματο με αυτά που εμεί υποστηρίζουμε ω Επιτροπή Προπολισμών και αυτό με εξέπληξε Ιδίω με κάποιε κυβερνήσει που δεν τι θεωρούσα και τόσο φιλοευρωπαϊκέ, ε, πάντω έδειξαν τη θέληση να συζητήσουν και για του ίδιου πόρου και για το επίπεδο του προσεχού ε, πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου, ότι αναγνώρισαν την ανάγκη να υπάρξουν νέοι πόροι λόγω των νέων προτεραιοτήτων. Άρα βγήκα πιο αισιόδοξα από την μπήκα στην αίθουσα. Και ιδίω όταν πήρα κάποιε πληροφορίε για το τι έγινε στα πάνελ το πρωί που μιλούσαν για τα ιατρικά ταμεία και την κοινή γεωργική πολιτική. Ότι είναι δύο σιρτάρια γεμάτα με χρήμα που θα μπορούσαν από αυτά να βγάλουν κάποια κονδύλια και να χρηματοδοτήσουν το μέλλον. Ε, σε σχέση με το πρώτο, το απογευματινό πάνελ ήταν πολύ ελπιδοφόρο. Ε, και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε γρήγορα να καταλήξουμε σε μια καλή συμφωνία που όπως είπατε πολύ σωστά κύριε Πρόεδρε από την πρώτη πρώτη στιγμή θα πρέπει σε αυτές τις διαδικασίες να συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να έχει το λόγο του. Για το προσεχές δημοσιονομικό πλαίσιο, κύριο Σόλμπριχτ. Ευχαριστώ. Είμαι ελαφρώς λιγότερο αισιόδοξο από την συνάδελφο. και οι υπουργοί είχαν πολύ συγκεκριμένε απόψει. Δυστυχώ δεν είχαμε από τους καθαρούς πληρωτέ ε, υπουργούς, γιατί θα τα βλέπαν αλλιώ τα πράγματα. Άρα ας προχωρήσουμε προς τα εκεί και όπως είπατε και εσείς. θέλουμε να υπάρχει σοβαρή συνεργασία. Και μιλάμε για συνεργασία με τους υπουργούς, με κάθε σεβασμό προς τους συνεργάτες υπαλλήλου. Θέλουμε, δεν λέμε για συνεργασία με εκείνους. Νομίζω ότι η επόμενη σύνοδος θα γίνει τον Ιανουάριο. Και αξίζει να πάει κανείς εκεί να δει τι γίνεται. Ε, η πρωινή σύνοδος για τη συνοχή δεν ήταν τόσο αισιόδοξη πάντως. Ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θέλω να έρθω σε ένα άλλο θέμα σημερινή ψηφοφορία. Το πρόβλημα είναι ότι η ψηφοφορία καθορίστηκε τελευταία στιγμή και αυτό είναι πρόβλημα για πολλούς συναδελφούς ε, για να μπορέσουν να έρθουν. Γιατί όλοι έχουμε, παρακολουθούμε τρεις-τέσσερις επιτροπές και πολλές άλλες δραστηριότητες στο Κοινοβούλιο. Εγώ σήμερα π.χ. το πρωί είχα μια συνάντηση στη Γενέβη του ΠΟΕ και επειδή άλλαξαν τα πράγματα δεν πήγα τελικά κάτι το οποίο κόστισε στο Κοινοβούλιο. Τα πράγματα αυτά πληρώθηκαν και οι συνεργάτες επίσης οι οποίοι τα είχαν προτεμάσει δεν μπορούν να πάνε στον ΠΟΕ γιατί τελευταία στιγμή ε, γίνεται ψηφοφορία. Έχω μια παράκληση ψηφοφορίες και αυτές εδώ είναι οι σημαντικότερες του έτους να προγραμματίζονται μακροπρόθεσμα και όλοι οι βουλευτές να ξέρουν πότε θα λάβουν χώρα. Ε, είναι νομίζω το ελάχιστο έτσι. Αλλιώς ε, έχουμε ανηλυμένες υποχρεώσεις που πρέπει να τις ακυρώσουμε γιατί δεν υπάρχει προγραμματισμός. Παρακαλώ λίγο στο μέλλον να προσαρμόζεται ο προγραμματισμός και στου βουλευτέ δεν έχουμε μόνο την Επιτροπή Προπολογισμού, αλλά έχουμε πολλές δραστηριότητες ε, εξίσου μεγάλη ε, σημασία. Αλλά βεβαίως η σημαντικότερη είναι η ψηφοφορία αυτή, είναι η σημαντικότερη ψηφοφορία του έτους, γι' αυτό αναγκάστηκα να ακυρώσω την άλλη μου υποχρέωση. Σας ευχαριστώ. Ναι, έλαβε αυτό το οποίο είπατε, διόντως ε, υπήρξε αυτή η δυσκολία. Όσον αφορά το να αποφασιστεί οριστικά το χρονοδιάγραμμα, η μέση διάταξη, αλλά όπως ξέρετε ε, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη για τον Σεπτέμβριο ε, θα είναι θεματικά αφιερωμένο σε αυτή τη δουλειά. Οπότε εδώ και δύο χρόνια αυτό κάνουμε. Να κλείσουμε συμβασμούς, να ε, χτενίσουμε τις προτάσεις του εισηγητή των σκιωδών, αλλά τελικά άρχισε η υπόθεση. Οπότε να προσέξουμε το χρόνο. Το χρονοδιάγραμμα, το, τα ωράρια, όλα αυτά να είναι από νωρίτερα γνωστά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σε όσα ήδη είπαμε για την περίοδο μετά το 2020 για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Προσθέσω τα εξή που αφορούν την Επιτροπή μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι πρόκειται περί ιστορικής ευκαιρίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τον προϋπολογισμό μας. Και Ε, κατόπιν των χθεσιών εξελίξεων είμαστε όλοι πάρα πολύ ικανοποιημένοι αλλά μην παραζηρώμεθα. Η μάχη στο Συμβούλιο θα είναι σκληρή. Ε, το, τα κουσούρια δύσκολα τα αποβάλλει κανείς. Οπότε και είναι καθήκον μας να κάνουμε ό,τι παίρνει από το χέρι μας. Και έτσι να αποκρισταλώσει το Κοινοβούλιο μια θέση ξεκάθαρη. Άλλη ευκαιρία δεν θα υπάρξει. Αυτό είναι το πνεύμα του κειμένου που τώρα εκπονώ για την Επιτροπή Δημιουργικού Ελέγχου. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Πρόεδρε, πρώτα σας διακόψω. Να ξεκαθαρίσουμε το εξής εγώ και η κυρία Γκάρτια Σάμπαλ, δεν συζητούσαμε ε, τέτοιες εντυπώσεις. Ε, ήταν θέμα ουσίας. Η ουσία έχει σημασία. Ήταν, υπήρχε κάποιο πραγματικό περιεχόμενο ή όχι. Έχετε δίκιο εδώ πέρα βεβαίω. Έχουμε αυτό το παράθυρο ευκαιρία και πρέπει να προσέχουμε, δηλαδή έχουμε μόνο θετικές παρατηρήσεις ή έχουμε κάποια ουσία. Η ανάλυση μας ήταν η εξή. Εμείς είδαμε τα πρώτα σημαδιά ουσία. π.χ. είχαμε μια σοβαρή συζήτηση ιδίων πόρων. Αυτά ήταν τα μηνύματα χτε. Και είναι κάτι το καινούριο. Αντιλαμβάνομαι αυτό το οποίο λέτε. Ε, γι' αυτό ακριβώς ε, θα ήθελα να εκφράσω την άποψή μου. Αυτό είναι λοιπόν αυτό το στοιχείο. Ευχαριστώ. Ναι, αλλά όσον αφορά αυτή την επιλογή για τους ίδιους αυτό θα σημαίνει ότι θα πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε για καθαρούς εισφορείς, ε, καθαρούς εισπράττοντες ας πούμε. Οπότε, τι θα γίνει με τις φιλοδοξίες μας. Έχουμε τι αποφάσει των ε, συντονιστών, καθώς κάποιε κάποιες ε, εκθέσεις, Γκάιερ, για τις ε, κοινωνικές για την ΛΥΜΠΕ, όσον αφορά τον κανονισμό της ΕΝΙΣΑ. Επίσης, για την κυβερνοασφάλεια, την κατάρριξη του σχετικού κανονισμού και την πιστοποίηση του ΕΛΚ για την Επιτροπή Ελίας για το πρωτόκολλο των ευκαιριών Ελίας Επίσης, αποφασίστηκαν από, τα θέματα για τα εργαστήρια και τις ακρόασεις. Για το 18 θα γίνει μια ακρόαση όσον αφορά την αξιολόγηση των ροών χρηματοδότηση που αφορούν την μετανάστευση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. επίση άλλη ακρόαση αποφασίζει και όσον αφορά τι εξωτερικέ απόψεις της μετανάστευσης, όσον αφορά επίση τα εξωτερικά καταπιστεύματα. Τρίτη ακρόαση, το μέλλον της προσπαρασκευαστική δράση όσον αφορά την έρευνα για την ε, άμυνα και επίση νέοι πόροι για την κοινή πολιτική άμυνα. Τέταρτο θέμα, ο προπολογισμό της Ένωση και Συμφωνία των Παρισίων για το κλίμα. Οι συντονιστές επίσης αποφάσισαν και για τις αποστολές που θα κάνουμε. Η πρώτη στην Ιρλανδία, την Πράσινη Εβδομάδα του Φεβρουαρίου. Μετά για την Πράσινη Εβδομάδα του Απριλίου θα ταξιδέψουμε στην Μορδαβία, τον Μάιο στην Ισπανία, στη χώρα των Βάσκων, για να δούμε τι γίνεται με την αξιοποίηση των ε, κοινωτικών κονδυλίων και τον Ιούνιο Ισραήλ-Παλαιστίνη. Η Επιτροπή των Προπολογισμών επίση το 2018 θερμοσύνει ένα εργαστήριο όσον αφορά τα δημοσιονομικά θέματα για την Ευρωζώνη. Πώ είναι η κατάσταση, πώ θα εξελιχθεί. Γιατί όλα τα κρατημέλη θέλουν να γίνουν μέλη της Ευρωζώνης. Ε, επίσης να έχουμε τέσσερις μελέτες που να προετοιμαστούν από την υπηρεσία για την πολιτική συνοχής, δεύτερη μελέτη για την επισήμανση το που έχουμε δαπάνες, που έχουμε επιστροφές από τους αποδέκτες και δικαιούχους των παροχών επίσης για τα υπόλοιπα προς ε, ανάλωση και χρηματοδότηση του προπολογισμού από πόρους πέραν των ιδίων πόρων. Φερρυπίν επιστροφές, Φερρυπίν από θεωρήσεις εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα σχετικά έσοδα πάνε στον προϋπολογισμό μας. Αυτά προς ενημέρωσή σας. Έχετε λάβει τα πρακτικά για τις προηγούμενες συναντήσεις μας. Έχετε κάποιες ε, παρατηρήσεις. Αν δεν υπάρχει κάποια ένσταση, εγκρίνονται τα πρακτικά. Και τώρα δούμε τι γίνεται για την κοινή προσπαθειά μας με την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου που αφορά τις εξελίξεις για τον τριμερή διάλογο ή τους τριμερείς διαλόγους που διεξάγονται ούτως ώστε να υπάρξει απλούστευση στην διαδικασία που αφορούν τον δημοσιονομικό κανονισμό. Να έχει την καλοσύνη να λέω το λόγο η ε, κυρία Γκρέσλε και κατόπιν ο συνεισηγητής ο κύριος Σφάρτς. Ακολουθεί η Πρόεδρος της Επιτροπής των Προϋπολογισμών. Όλα αυτά, όσες προσπαθίες σας έχουν εκδημηθεί σε όλες τις χώρες. Να, επομένως, πόσο παιδαγωγικές είναι αυτές οι αποστολές που κάνουμε. Γκρέσλε. Σε τα καλά σας λόγια, αλλά είναι δική περίπτωση αυτά. Ναι, τρίτη συνεδρίαση, πάλι τέσσερις ώρες, διατρέξαμε 40 άρθρα ε, μέχρι την σελίδα 283 και απερίψαμε τα, 67, τα 64 μέχρι 67 τα άρθρα για τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ΣΔΙΤ και τις γενικές ε, διατάξεις για τους ε, χρηματοπιστωτικούς ε, δρόντες. Δεν είπαμε τίποτα τώρα για την διαχείριση των κοντιλίων εδώ πέρα, ειδικά την συνεργασία με την ΕΠΟ, Εθνικές Εξηγήσεις και τη χρηματοδότηση του ΕΦΣΙ για τους ενιαίους κανόνες Έχουμε ένα συνδυασμό διαφόρων προγραμμάτων και εκεί πέρα επίσης δεν καταλήξαμε σε κάποια συμφωνία. Ε, στο ερώτημα δηλαδή ποιος επιτρέπεται να ιδρύει ε, ευρωπαϊκές υπηρεσίες και εκεί πέρα δεν καταλήξαμε κάπου και υπάρχει βέβαια και το θέμα των αποκεντρωμένων και εκτελεστικών υπηρεσιών ε, και για τον εξωτερικό έλεγχό τους. Μετά αφήσαμε και το άρθρο 73 ανοιχτό το οποίο αφορά την απόδοση. Η απόδοση είναι πάρα πολύ σημαντική βεβαίως και πρέπει να λαμβάνετε υπόψη στην αξιολόγηση των προγραμμάτων. Κάτι επίσης το οποίο αφορά πολλά, προγρα... πολλά άρθρα αφορά ακριβώς το πάνελ διοικητικών ποινών. Η επόμενη συνεδρία είναι την 5 του Στρασβούργου και θα ξαναρχίσουμε από την αρχή γιατί έχουμε πολλά ανοιχτά σημεία για τα άρθρα 1 έως 84 για να τα θυμόμαστε. Μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου έχουμε άλλες δύο συναντήσεις και δύο επιπρόσθετες ε, συναντήσεις αρχές Νοεμβρίου. Και δυστυχώς ε, υπάρχει και μια συνάντηση που πρέπει να αναβληθεί λόγω σύγκρουσης με άλλη ε, σύμπτωση. Και έχουμε λοιπόν κάποια πράγματα, αλλά εντάξει τουλάχιστον προχωράμε. Uh, Ευχαριστώ, ο κύριος Ashworth. Δεν έχω να προσθέσω και πολλά σε σχέση με όσα είπε η συνεισηγήτρια. Θέλω απλά να σας υπενθυμίσω ότι ουσιαστικά θέλαμε να έχει ολοκληρωθεί στα τέλη οκτω... ε, συγγνώμη, φθινοπόρου το κείμενο αυτό. 12 ώρες μέχρι στιγμή έχει διαρκέσει ο τριμής διάλογο. Ούτε δεν έχουμε ε, διατρέξει το μισό κείμενο για πρώτη φορά. Και υπάρχουν σημαντικοί τομεί που τα θεσμικά όργανα διαφωνούν και θα πρέπει να γίνει πολλή δουλειά. Παραλαμβάνω ότι δεν έχουμε καν δει και πολύ μεγάλο μέρος του κειμένου για, καν για την πρώτη φορά. Είναι αδύνατον να έχουμε ολοκληρώσει μέχρι το φθινόπωρο που ήταν το αρχικό χρονοδιάγραμμα Ήδη όμω έχει καταβληθεί σημαντική προσπάθεια, πολλή δουλειά έχουμε κάνει. Θέλω να ευχαριστήσω τη συνεισηγήτρια και εσάς κύριε Πρόεδρε που ήσασταν πολύ συνεργάσιμο, υποστηρικτικό και ελπίζω την επόμενη εβδομάδα να σημειώσουμε λίγο περισσότερη πρόοδο. Ευχαριστώ πρόεδρο. Ωραία. Σα ευχαριστώ. Μπορούμε να ολοκληρώσουμε εδώ αυτή την ενημέρωση εκτό αν οι σκιώδεις θέλω να μα αναφέρουν τι δικέ του απόψει. Δεν θέλουν. Περνάμε λοιπόν στο επόμενο σήμα τη διάταξη. Ευχαριστώ την ε, κυρία Κράση και τον κύριο Άσχορθ. Και θα δώσω το λόγο τώρα στην Μόνικα Χολμάγερ που θα μας μιλήσει για την πολιτική την κτηριακή. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα μόνο μια σύντομη πληροφορία πριν περάσουμε στις ε, ψηφοφορίες και τις αποφάσεις. Υπάρχει ένα έργο κτηριακό που έχει ανακοινωθεί και δεν έχουμε καμία νεότερη πληροφορία. Είναι το Γραφείο Πληροφόρησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της ε, Κομισιόν ε, εις ε, Παρισίους. Άνοιξη του 2018 υποτίθεται ότι θα γίνει η μετακόμιση σε ένα νέο κτίριο το οποίο είναι φτηνό για τα δεδομένα του Παρισιού οι αιτίε μετακόμισης είναι λόγια ασφαλείας, ε, το ότι δεν υπάρχει επαρκής χώρος για εκδηλώσεις, ε, επίσης απαιτούνται δομικές ε, ανακαινήσεις και δεν μπορούσαμε επίσης να βρούμε κάτι το οποίο θα, στο οποίο θα μπορούσαμε να πούμε πριν εκπνεύσει η τωρινή συμφωνία ενοικίασης που έχουμε. Αυτά έχουμε λοιπόν ως πληροφορίες. Ε, θα υπάρξουν και άλλες που θα μας αποστείλουν λεπτομερέστερες μόλις υπάρχουν περισσότερα δεδομένα. Σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Πώς προχωρά το θέμα. Και φαντάζομαι θα μας ενημερώσουν να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για την ε, Μετακίνηση λοιπόν της Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας στο Παρίσι κτίριο υπάρχουν ερωτήσει. Αν όχι να περάσουμε στις ψηφοφορίες. Βάλτε τις κάρτες σας παρακαλώ στο μηχάνημα. De vote électronique pour vérifier euh, que tout fonctionne parfaitement. Για να δούμε κατά πόσον λειτουργεί το σύστημα. Άρχεται η ψηφοφορία. Η Δοκιμαστική. Έχουμε 31 δυνητικούς ε, ψηφίζοντες. 33. 34. Ah, 34. 35. 35. Δεν έχει την κάρτα του ο Γενικός Εισηγητής. Θα μας τα λέει κάθε φορά. Λοιπόν, 36 ψηφίσαντες και οι τρεις από αυτούς που έχουν κάρτες δεν έχουν ψηφίσει. Ένας είμαι εγώ από τους τρεις. Εντάξει, πάει ο ένας. Λοιπόν, πέρας ψηφοφορίας, δύο ψήφοι. Λοιπόν, δεν πειράζει. Τμήμα 3. Κύριε Γκάγερ, έχουμε κάποιο αίτημα για κάποια μεταφορά πίστοσης. Όχι. Για τα άλλα τμήματα, αυτό είναι το τμήμα 3, ο κύριος Τάραντ, για τα υπόλοιπα τμήματα πλήν του τμήματος 3, κύριε Τάραντ. Um, thank you, Mr. Uh, Ευχαριστώ. Για να ξεκονομήσουμε χρόνο, δεν θα αναλύσω αυτά τα οποία μπορείτε να διαβάσετε στους φακέλους σας. Έχω συζητήσει με όσους έχουν κάνει τα αιτήματα και παρά το ότι επιφυλακτικός επίστην. Pour la synthèse très, très Περνάμε λοιπόν σε μάλλον στι επόμενε προφορίες γιατί θα θεωρήσουμε ότι οι τέσσερις αυτές μεταφορές μεταφορέ πιστώσεων χρειάζεται να ψηφιστούν, γίνονται δεκτές και η τροποποίηση του οργανογράμματος επίσης γίνεται δεκτή. Εκτός αν κάποιος θέλει να ψηφίσουν παρόλα αυτά. Αν όχι, θεωρώ ότι εγκρίνει η Επιτροπή τι μεταφορέ πιστώσεων και την αλλαγή του οργανογράμματος. Και περνάμε στην κτηριακή πολιτική. Θα ξαναδώσω το λόγο στη Μόνικα Χολμάγερ για να μας παρουσιάσει την άποψή της και μετά θα περάσουμε στην ψηφοφορία. Also, an Anfang stelle ich ganz kurz... Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα υπάρχει ένα έργο της Κομισιόν στο Λουξεμβούργο που θέλουμε να αναπληθεί για δύο εβδομάδες για να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις. Πρόκειται για ένα κτίριο που προκύπτει από το πρόβλημα του ότι το κτίριο Ζαν Μονέ ε, λόγω του 2014 έπρεπε να εγκαταληφθεί επιγόντως λόγω αμοιάντου και επιπλέον ε, νοικιάσαμε κάποια άλλα κτίρια για μια μεταβατική περίοδο στην πτέρυγα 2 του κτηρίου Ντρόσμπαχ ε, και αλλού και η κατάσταση στο Ζαν Μονέ ήταν ότι είχαμε 7.000 ε, τετραγωνικά μέτρα κυρίως αποθηκευτικούς χώρους. Προβλήματα τα οποία υπήρχαμε με την πεταπατική κατάσταση είχαμε ε, πάνω από 1500 τετραγωνικά μέτρα δεν έφταναν, έπρεπε ε, διάφορα γραφεία να εγκαταληφθούν οι εργασίες πήγαιναν πάρα πολύ αργά και ε, υπήρξαν κάποιες συμβάσεις επίσης που απορρίφθησαν. Επίσης έχω κάποιες ερωτήσεις για την Κομισιόν και θα ήθελα να αναβληθεί μέχρι την επόμενη συνεδρίασή μας γιατί έχουμε και ένα κοντέινερ όπου δεν είναι προσβάσιμα τα αντικείμενα, το νίκιο είναι 6.500 ευρώ το μήνα, αλλά υπάρχουν πράγματα, ε, παραδείγματο χάρη το προσωπικό της αρμόδιας γενικής διεύθυνσης για λόγους αστικής ευθύνης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει το υλικό του Κοινοβουλίου. Ε, δεν είναι δυνατόν να αγοράζουμε όμω τα πράγματα δύο φορέ. Πρέπει να αλλάξουν οι σχετικοί κανόνε. Γιατί, δηλαδή, τι πρόβλημα υπάρχει μεταξύ δύο θεσμικών οργάνων και δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον εξοπλισμό ένα του άλλου. Και μετά. Οι διατάξει Κομισιόν ε, λένε ότι δεν μπορεί να υπάρχει εσωτερικό και εξωτερικό προσωπικό στον ίδιο χώρο και έτσι εξηγείται η ανάγκη ενοικίασης ε, νέων χώρων. Επίσης υπάρχει αυξημένο κόστος ε, μεταφοράς για το προσωπικό. Αλλά τώρα θέλουν να νοικιάσουν νέο κτίριο, αλλά η ε, νέο κομμάτι του κτηρίου, αλλά είναι μεγαλύτερο το νίκιο για το συγκεκριμένο τμήμα του κτιρίου από ό,τι για το υπόλοιπο. Επίση θα μπορούσαν να υπολογίσουν μόνο το κόστος ενοικίου και όχι μετασκευής, αλλά κατ' ουσίαν αν βάλουμε και τη μετασκευή μιλάμε για διπλασιασμό του ενοικίου και θέλω να το συζητήσω αυτό με την Κομισιόν. Γι' αυτό ζητάω αναβολή για δύο εβδομάδες ε, και προτείνω να περιμένουμε πως η Κομισιόν ε, δώσει ικανοποιητικές ε, απαντήσεις. Αλλά θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και για την αντίθετη περίπτωση γιατί διπλάσια τιμή για τέσσερα χρόνια που είναι η μεταβατική περίοδος μέχρι να είναι έτοιμο το επόμενο κτίριο είναι πολύ. Δεύτερον, το δεύτερο κτίριο δηλαδή της Κομισιόν δεν έχει κανένα πρόβλημα, είναι το κτίριο CDMA και Β28 το ΕΝ ξεκίνησε το 2004. Εκεί σε αντίθεση με το άλλο τα πράγματα είναι πολύ θετικά. 5,9 εκατομμύρια και 4,3 εκατομμύρια θα δώσουμε στα δύο κτίρια αυτά. Ε, και 26% λιγότερο και στο άλλο κτίριο έχουμε πάει από τα 4,1 στα 3,1 εκατομμύρια ευρώ μείον 24% δηλαδή κάτι το οποίο βεβαίως ε, σημαίνει σημαντική και αποτελεσματική μείωση του κόστους και σας παρακαλώ αυτά τα δύο κτίρια να τα εγκρίνετε. Ερωτήσεις, παρατηρήσεις για το κτίριο, για το κτίριο στο Λουξεμβούργο. Αναβάλουμε για δύο εβδομάδες και για τις Ρυξέλλες, στην οδό Σάντε Μάρς, πεδίου του Άριος και στη Ριμπελιάρ για τα κτίρια. Η συγγήτρα είναι υπέρ. Εφόσον θα συνιστά αυτό οικονομία, εξοικονόμηση. Λοιπόν, διανατάσσω στις χειρός. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν. Examen et plutôt vote des amendements. Ψηφίζουμε τώρα τις τροπολογίες για τον περιβολισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2018. Πολύ σημαντική, το είπα και στην αρχή, και η σημερινή και η αυριανή συνεδρίαση, γιατί δεν νομίζω θα ολοκληρώσουμε σήμερα και θα χρειαστεί να συνεχίσουμε και αύριο το πρωί. Διότι πρέπει να ψηφίσουμε 2.392 τροπολογίες που έχουν κατατεθεί για το σχέδιο προπολογισμού του 2018 από την Επιτροπή, από τις ομάδες και από τους ηγητές. Ζίγκφριτ Μούρεσαν και Ρίτσαρντ Άσχουερθ δούλεψαν εντατικά. Θέλω να τους ευχαριστήσω, να τους συγχαρώ. Ηράκλειον το έργο που ανέλαβαν εδώ και μήνες να φέρουν σε πέρας. Κατατέθηκαν πολλά ψηφίσματα και έγγραφα εργασία και την τελευταία εβδομάδα είχαμε και την εξέταση των τροπολογιών και την εκπόνηση συμβιβαστικών προτάσεων. Πολύ δύσκολη δουλειά. Αν λοιπόν συμφωνείτε μπορούμε να περάσουμε στην ψηφοφόρια. Σήμερα θα ψηφίσουμε τις τροπολογίες μας στο τμήμα 3, προϋπολογισμός της Επιτροπής, κατηγορία 5, διοικητικά, διοικητικές γραμμές και οργανισμοί. Μετά, κατηγορία 1α, 1β, 2, 3, 4, έσοδα και δικά μέσα αν προλάβουμε, μπορεί να ψηφίσουμε και τα πιλωτικά και τις προπασκευαστικές. Και έχοντας υπόψη μας ότι πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει 6 και μισή. Θα ολοκληρώσουμε αύριο την ψήφα οφορία από το τμήμα με ό,τι δεν έχει ψηφιστεί σήμερα. Μετά πληρωμές, μετά τα υπόλοιπα τμήματα. Και θα ολοκληρώσουμε με το τμήμα 1 που είναι ο προπολογισμό του Κοινοβουλίου. Πριν ψηφίσουμε όμω, θέλω να δώσω το λόγο στου ηγητέ μα για να μα πούν ποια είναι η δική του προσέγγιση και ποιο είναι το πνεύμα που του ε, καθοδήγησε στι συμβασικέ προτάσει που έχουν καταθέσει. Ο Ζίκφριτ Μούρεσαν πρώτα απ' όλα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κάλλιες, πέρα συναδελφοί, πρώτα πρώτα ευχαριστίες προς όλους τους συναδελφούς που εντατικά συνεργάστηκαν τις τελευταίες εβδομάδες. Οι ισχυώδες, ε, οι πολιτικές ομάδες, οι συνεργάτες, οι υπάλληλοι των πολιτικών ομάδων, η γραμματέα μας βέβαια, όλοι αυτοί ήταν ε, κορυφαία σημασία στο σώστο. σήμερα να μπορέσουμε να έχουμε αυτή την δέσμη προτάσεων που νομίζω ότι είναι στο ίδιο μήκο κύματο με τι προτεραιότητε του Κοινοβουλίου, όπω διατυπώθηκαν σε αρχέ εναστότω έτου και επίση είναι στο ύψο των προσδοκιών που τρέφουν οι Ευρωπαίοι, ε, ε, Ευρωπαϊκέ, ε, ή μάλλον από μεριά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να δούμε τι έχει αυτό το πακέτο συμβασμών. Πρώτα-πρώτα θέλουμε να επικαλεστούμε τι διατάξει τη ευελιξία του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου, ούτω ώστε να καλύψουμε τι πολιτικέ προτεραιότητε όπω προείπα πρώτα-πρώτα. Βέβαια, απορρίπτουμε όλε τι περικοπέ του προπολισμού που είχε προτείνει το Συμβουλίο, γιατί θεωρούμε ότι εάν δεχτούμε αυτέ τι περικοπέ του Συμβουλίου που προβλέπουν λιγότερου πόρου για έρευνα, καινοτομία, υποδομέ, μικρομεσαίε επιχειρήσει ακριβώ του τομεί εκείνου που ισχυροποιούν την Ευρώπη και εάν το δεχτούμε όλα αυτά, ε, τότε αυτό θα είναι ένας κατήφορος για πιο αδύνατη ένωση, πιο αδύνατο προϋπολογισμό. Ε, για αυτό ακριβώς και εμείς θέλουμε να μην επέλθει, μην έρθει και μην γίνει καμία περικοπή. Όλθα θα είναι Να, πρόκειται για ακριβώς ότι τις, τους πόρους που χρειάζονται ένα σωρό έργα και σχέδια. Επίσης, έχει προτείνει η Κομισιόν το να υπάρχει μια, μια θεσμική ρύθμιση για αλληλεγγύη. Συνεχίζεται η σχετική νομοπαρασκευαστική διαδικασία. Είναι αξιόλογο αυτό το όραμα, αλλά δεν μπορούμε να προδικάσουμε την κατάληξη της ιστορίας. Γι' αυτό και πάμε να μην γίνουν περικοπές στα κονδύλια εκείνα τα οποία πρόκειτο να, αυτό το, το σώμα, τέλος το φορέα ελεγγύης να τον ε, πρικοδοτήσουν. Επίσης, έχουμε και όλες τις περικοπές για το ΕΦΣΙ, για το Μισοτικών Επενδύσεων. Δεν θέλουμε να γίνουν ούτε αυτές τις περικοπές. Έχουμε επίση το κεφάλαιο 1α μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Εκεί έχουμε προτείνει αυξήσει 143 εκατομμυρίων. Και επίση το περιθώριο είναι 5-6 εκατομμύρια. Μας ενδιαφέρουν οι θέρμα να από τα χρήματα στις ΜΜΕ. 22 ε, για το κόσμο, 15 για το Συμβούλιο Έρευνας και 10 για το Marie Curie και 32 ε, εκατομμύρια για το έρασμος αλλά και άλλα 8 για ε, ειδικά ειδικέ ετήσιες εκδηλώσει. Ε, ε, ε Επίση, συνεργαστήκαμε, τα βρήκαμε τι πολιτικές ομάδες τις υπόλοιπε για την πρωτοβουλία που αφορά την ανεργία των νέων που ήδη μαστεί στην Ευρώπη και θα έχουμε εκεί 253 εκατομμύρια όπω θα προτείνει η Κομισιόν. Όμως αυτά τα 233 είναι φραγκοδίφραγκα σε σχέση με αυτά που χρειάζεται η Ευρώπη για να αντιμετωπίσει την ε, ανεργία. Οπότε είπαμε οι πολιτικές ομάδες να ζητήσουμε 600 εκατομμύρια για αυτή την πρωτοβουλία του νέου του χρόνου. Δεύτερο κεφάλαιο θέλουμε να έχουμε περιορισμένες ε, αυξήσεις, ιδίως όσον αφορά τα θέματα για το κλίμα, 21 εκατομμύρια και άλλα 6 εκατομμύρια για γαλακτοκομικό τομέα και την αποθεματοποίηση, όπως είπε η Επιτροπή Γεωργίας, και άλλα 50 εκατομμύρια για τους νέους γεωργούς. Πολύ σημαντικό, γιατί θέλουμε οι νέοι να έχουν περισσότερες ευκαιρίες και στα θέματα γεωργίας. Γιατί αυτά τα χρήματα για τους νέους ε, γεωργούς σημαίνει περισσότερη επασχόληση Τώρα μετανάστευση και ασφάλεια ε, να αντιμετωπίσουμε το προσφυγικό είναι μία από τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου και για αυτό και επίσης προσέχουμε τι θα κάνουμε για το κεφάλαιο 3. Όπως ξέρετε και εδώ υπήρχε 0, μηδενικό περιθώριο. Να ενισχύσουμε, είπαμε, τις ε, κοινωτικές αποκεντρούμενες ε, υπηρεσίες γιατί θα πρέπει να εκταμιεύσουμε περισσότερους πόρους για αυτές τις υπηρεσίες εκεί όπου χρειάζεται να έχουν περισσότερες αρμοδιότητες, να κάνουν περισσότερα αλλά να μην δαπανίσουν και πάρα πολλά. Europol 10 εκατομμύρια, Εάζο 26 ΣΕΠΟΛ 3,3, Eurojust 3,1 εκατομμύρια ευρώ και τώρα για να δώσουμε το, το, να στείλουμε το μήνυμα ότι συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε το προσφυγικό, το μεταναστευτικό, αυξάνουμε στο ΑΜΙΦ τη χρηματοδότηση κατά 20 εκατομμύρια και για το Ταμείο Ασφάλειας κατά 50 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, αλλά 21 εκατομμύρια θα θέσουμε για πολιτιστικά και θέματα των πολιτών. Όπω γνωρίζετε συναδελφοί, θα πρέπει ακόμα να αποφασίσουμε το πολύ σημαντικό τι θα γίνει για το μέσο διευκόλυνση, δηλαδή του πόρου προ την Τουρκία. Αυτό εκκρεμεί, ακόμα δεν έχει κλείσει. Όσο και αν είναι αβέβαια πράγμα, να μην συνεχίζουμε τι προσπαθίε μα με υπεύθυνο τρόπο. Δεν θέλουμε να υπερβούμε το περιθώριο του κεφαλαίου 4 και προτείνουμε αυξήσει κατά 120 εκατομμύρια όσον αφορά την πολιτική νοτιογειτονία γιατί εκεί, εκεί είναι μεγαλύτερη πίεση, εκεί είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα. 25 εκατομμύρια για πολιτική γειτονία προ Ανατολά και 35 για Βαλκάνια ούτως ώστε να βοηθήσουμε να υπάρχει περισσότερη σταθερότητα στην περιοχή ε, και διάφορα προγράμματα για το Erasmus στο 426, 22 για την τουρκοκυπριανική κοινότητα. Αυτό είναι σημαντική βοήθεια του προπολογισμού, Όσον αφορά το κυπριακό, 28 εκατομμύρια για ανθρωπιστική βοήθεια επίσης. Και συζητήσαμε, οι συγητές, είναι οι τι θα γίνει για τη χρηματοδότηση της Τουρκίας. Οπότε και αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε τη γνώμη των εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής Εξωτερικών και να είμαστε στο μήκο κύματο ε, του να βοηθήσουμε τις πολιτικές μεταρρυθμίσεις στη χώρα. Να γίνουν κάποιες περικοπές λόγω των ε, εκεί εξελίξεων. Δεν πιστεύουμε ότι τώρα η Τουρκία βρίσκεται στο δρόμο των πολιτικών μεταρρυθμίσεων σε ευρωπαϊκά πρότυπα. Ε, γι' αυτό και αποφασίσαμε να περικόψουμε το κονδύλι κατά 50 εκατομμύρια και να δώσουμε 30 εκατομμύρια στο αποθεματικό διότι θέλουμε να αλλάξει η Τουρκία. Θέλουμε θετικές πολιτικές εξέλιξεις Γι' αυτό και τα χρήματα πάνε στο αποθεματικό. Να το μείνουμε, θα στείλουμε. Θα του τα δώσουμε τα λεφτά, άπαξ και η ελευθερία του λόγου, ανθρωπινό δικαίωμα, δικαιώματα, θεμελιώδης ελευθερία και πάλι πρετανεύσουν στην χώρα. Ε, επίσης, επίσης, για τις άλλες αποκεντρωμένες υπηρεσίες προτείνουμε πέραν των θεμάτων δικαιοσύνης, υπηρεσιών δικαιοσύνης δηλαδή και ιστορικών, ελαφρές, ελαφρές. Αυξήσεις 5,5 για την ΕΑΣΑ λόγω της νέας νομοθεσίας γιατί υπάρχουν εξημένε αρμοδιότητε τώρα για την υπηρεσία αυτή. Αυτή μια γενική έποψη ανά κεφάλαιο, Πρόεδρε. Όμω τώρα χρειάζεται ξεκάθαρη εντολή από το Κοινοβούλιο. Σήμερα από την Επιτροπή μας και τέλος Οκτωβρίου από την Ολομελητός, ώστε να μπορούμε να έχουμε ισχυρές διαπραγματεύσεις, ισχυρά του στα χέρια μας για τις διαπραγματεύσεις τέλος πάντων και πρόκειται για το πακέτο που αποτελεί τις προτεραιότητες των ε, πολιτικών ομάδων, αυτά τα οποία θα είναι η γραμμή του Κοινοβουλίου. Οπότε, να, εν αναμονή της ψηφοφορίας, να σας ευχαριστώ για τη συνεργασία. Ξέρω ότι είναι σκληρή η δουλειά, αλλά νομίζω ότι καλά τα πήγαμε. Σας ευχαριστώ κύριε Γενική Συγητά. Και εσείς Κάνατε πάρα πολύ δουλειά και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ επίσης που μας διαφωτίσατε σε σχέση με τις ψηφοφορίες που θα ξεκινήσουν σε λίγο. Κύριε Άσχουεθ τώρα για τα λοιπά τμήματα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους της Επιτροπής, ε, τους σχεώδης ηγητές ε, και το προσωπικό για τη δουλειά που έκαναν και το πνεύμα συμβιβασμού που επέδειξαν. Και να υπενθυμίσω ότι ποτέ δεν είναι δύσκολο βεβαίω να βρεθεί η σωστή ισορροπία. Και ως αφετηρία να σας μεθυμίσω ότι φέτος τον Απρίλιο το Κοινοβούλιο είχε α, ορίσει την αύξηση του προπολογισμού μας στο 2,3% έχοντας κατά νου το επίπεδο του πληθωρισμού, θεωρούσα ότι είναι μια υπεύθυνη και λογική θέση. Γι' αυτό πρότεινα στην Επιτροπή μας να τεθεί αυτός μέτρο σύγκρισης για τα άλλα θεσμικά όργανα. Του του λεχθέντος όμως ανέφερα τρία θεσμικά όργανα τα οποία έχουν επιπρόσθετες απαιτήσει που είναι δικαιολογημένε και αναγκαίες και άρα ε, πρότεινα αύξηση πάνω από το 2,3%. Συγκεκριμένα το ΔΕΚ, το δικαστήριο που υπάρχουν αυξημένε απαιτήσει ασφαλείας και τη χρηματοδότηση της μετάφρασης. Και για το θέμα της, ε, εξωτερικής υπηρεσίας, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης απάντησα σε μια προτεραιότητα του Κοινοβουλίου που ήταν να υπάρξει μια ε, ομάδα στρατηγικής επικοινωνίας. Οι προτάσεις μου από την άλλη προσπάθησαν να υπάρξει μια δημοσιονομική πειθαρχία, δηλαδή κάνοντας οικονομίες αλλού να επιτύχουμε τον στόχο του 2,3%. Αυτό πρότεινα λοιπόν ένα πάγωμα σε δύο περιπτώσεις και στο... στην περίπτωση του ελεγκτικού συνεδρίου πρότεινα και εξοικονομήσεις. Μια που είμαι στο θέμα του ελεγκτικού συνεδρίου, να αναφέρω ότι υπάρχει ένα λάθος εδώ στον κατάλογο των ψηφοφοριών και θα ψηφίσουμε άπαξ για την ε, τροπολογία για τα επιπρόσθετα 3 εκατομμύρια στο αποθεματικό. Επίσης, να αναφέρω ότι έχω επιλέξει να ακολουθήσω το παραδοσιακό πρωτόκολλο και σεβάστηκα την λεγόμενη συμφωνία κυρίων και δεν προσπάθησα άρα να τροποποιήσω ή να μειώσω τον προπολογισμό του Συμβουλίου. Προστάτευσα επίσης από περικοπές τον συνήγορο του πολίτη και ε, αποκατέστησα τον προϋπολογισμό της, ε, του επόπτη προσωπικών δεδομένων. Τέλος, να τονίσω ότι οι προτάσεις μου είναι αποτέλεσμα συμβιβασμού. Στο μέτρο του δυνατού δέχτηκα τις προτάσεις άλλων ομάδων και επιτροπών. Και άρα θα ήθελα να τους ευχαριστήσω και πάλι για το πνεύμα που επέδειξαν και ελπίζω και προτείνω να είναι αυτή η πρόταση μια πρόταση υπεύθυνη που θα την στηρίξουν όλοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε εισηγητά. Ευχαριστούμε και τους και εισηγητές, όλους για τη δουλειά σας. Διότι έτσι είμαστε στη τώρα πια να ψηφίσουμε έχοντας γνώση των πραγμάτων. Οπότε, άρχεται η ψηφοφορία, ή μάλλον η ψηφοφορία. Ξεκινούμε από το τμήμα υπαριθμών 3 που αφορά το κονδύλιο 5 για τον προϋπολογισμό της Επιτροπής. Έχουμε δύο υποομάδες πρώτα-πρώτα για το Παράδειγμα παραδείγμα ένα υπέρ. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Κατά ε, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερη η και αφορά το παράρτημα πίνακας 2. Υπέρ, κατά. Α, αποχές. εγκρίνεται. Και τώρα. Τις χωριστές ψηφοφορίε. Πρώτα απ' όλα, Όλαφ. Πρώτη ψηφοφορία. 24, 01, 08. Υπέρ, κατά. Επαλήθευση, ηλεκτρονική. Ψηφίζουμε. Vous avez tous voté. Ψήφισαν όλοι, όχι από ό,τι φαίνεται, δύο από ό,τι φαίνεται δεν έχουν ψηφίσει. Εγώ πάντως ψήφισα. Bon, eh bien, Πέρα Και εγκρίνεται 21-13 και δύο εποχές. Και τώρα. Τα ε, αποθεματικά. Πρώτον, Όλαφ. Υπέρ. Κατά αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο θεματικό που αφορά τους μισθούς των μελών της Επιτροπής. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτωται, αλλά θα κάνουμε επαλήθευση ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε. Σκριτά εκλού. C'est repoussé. Απορρίπτεται. Άλλο αποθεματικό που αφορά τους ειδικού συμβούλους. Υπέρ, κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τρεις παρατηρήσεις. Πρώτη. 04-01-04-02. Και κόντρ. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερη παρατήρηση. Αφορά του ε, Ευρωπαϊκού Δημοσίου χώρου. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τρίτη παρατήρηση. 25.01.02.13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτωται. Nous en venons aux agences κοινοτικέ αποκεντρωμένε υπηρεσίε. Τρει υπομάδε. Πρώτα πρώτα. Έχουμε παράρτημα πίναξ 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερη υπομάδα. Παράρτημα πίναξ 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τρίτη ομάδα. Παράρτημα πίναξη 3. Υπέρ. Κατά. Αποχέα συγκρίνεται. Τώρα, χωριστέ ψηφοφορίε. Έχουμε μια σειρά τροπολογιών. 20. Ξεκινούμε από το 11 μέχρι το 040314. Pour objet, soit de Αφορούν είτε κάποιων κονδυλίων ή αφορά κάποια μείωση των πιστώσεων. Ε, λέει όχι ο εισηγητή για αυτέ. Τι λέτε, να ψηφίσουμε όλε μαζί αυτέ τι 20 τροπολογίε. Κανεί δεν ενίσταται. Ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι θέλουν να εγκριθούν αυτέ τι τροπολογίε. Όλε μαζί, όλε μαζί. Απεφασίστε, θα τους ψήφουμε όλες μαζί. Να σηκώσω τον κύριο είναι υπέρ αυτών των τροπολογιών. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Και εν λογοτροπολογίες απορρίπτονται. Και τώρα έχουμε τις παρατηρήσεις. Η πρώτη. Δεν επιδέχεται ψηφορία. Η δεύτερη, η 3302 07 αφορά το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Ισότητα των Φύλων. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 33-03-04 Η Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνδρομής Ποιοι είναι υπέρ Eurojust Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται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 Πρώτη υπομάδα τροπολογιών που επαναφέρει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερη υπομάδα που αφορά αυτό το σώμα την υπηρεσία τέλο πάντων αλληλεγγύης δεύτερος πίναξ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτη υπόμονα. Τρίτος πίναξ. Υπέρ. Κατά. αποχές εγκρίνεται. Τέταρτη. Πέραν του σχεδίου προϋπολογισμού τώρα. Ε, πίναξ Τέσσερα. Υπέρ. Κατά. αποχές εγκρίνεται. Πέμπτη υπομάδα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Nous en venons au vote euh, séparé. Nous avons euh, une série d'amendements qui vont de la Έχουμε τώρα όλες αυτές τις τροπολογίες. Ξεκινούμε από την 010405 και τελειώνουμε στο 0403 0107 οι οποίες αποτελούν αντικείμενο ψηφοφορίας όλες μαζί, για να δεν έχετε ένσταση. Ποιοι είναι υπέρ του να εγκριθούν όλες αυτές οι τροπολογίες. Ποιοι είναι κατά. Ποιοι απέχουν. Άρα απορρίπτονται. Τώρα. Μια συμβαστική τροπολογία. για το, την υποομάδα 4. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Επομένως, απορρίπτεται η τροπολογία Γκουε. Παρακάτω. Για την κατάργηση κονδυλίου υπέρ κατά αποχές. L'amendement est repoussé. Et vient à la ligne 0204 020 για την ε, υπομάδα 3 υπέρ κατά και αποχές. Εγκρίνεται. Γκουε. Καταπίπτει η τροπολογία. 04-03-01. 01. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτω. Κατόπιν οι τέσσερις επόμενες τροπολογίες που αφορούν το 04, 03, 01, 04, 07. Όλες μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 04, 03, 01 για την υποομάδα 1 συμβαστική υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Και κατά πολιτισμού 04, 02, 03 μικροχρηματοδότηση κοινωνικής επιχειρηματικότητας υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 08-02-03-01. Συμβαστική για υποομάδα 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Γκουε. Καταπίπτει τροπολογία 733. 08-02-03-02. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Καταπίπτει το 7034 η τροπολογία της ΓΚΟΕ. 080206 συμβιβαστική για την υποομάδα 3. Επαναφέρει τα επίπεδα χρηματοδότησης προ εύση, υπέρ, κατά αποχές. Εγκρίνεται. 7035 τροπολογία καταπίπτει. Ενέργεια σύνδεξης γιουρατών. 08, 03, 01, 01 υπέρ Αποχές απορρίπτεται η τροπολογία. Ε, υπό ομάδα 1, 12-02-01, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και η τροπολογία γκουε καταπίπτει. 12. κάτω από το σχέδιο προπολισμού υπέρ κατά Αποχές. Νομίζω απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται 23-13. 14-04-01. Συμβιβαστική υπόμαδα 1. Παναφορά πιστώσεων υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία Γκουε καταπίπτει. 15.02.02 Όλα μαζί τα θέματα εδώ. Μαζί με την 15.02.03 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτονται. 18.05.03.01 Συμβαστική υπομάδα 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία γκουε καταπίπτει. Κατόπιν, τα νέα κονδύλια που θεσπίζονται, τα οποία όμως επιδέχονται μια ομαδική ψηφοφορία από το 010206 στο 240252. Αν δεν υπάρχει ένσταση να τα ψηφίζουμε όλα μαζί. Ποιοι είναι υπέρ όλων αυτών των ε, κονδυλίων να σηκώσουν το χέρι κατά και οι αποχές απορρίπτονται αποθεματικά 12 με 2 με 3 δύο τροπολογίες των πράσινων 84-92 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται έκον 66-29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται παρατηρήσεις 020201 με πρώτη τροπολογία που αλλάζει ο τίτλος του κονδυλίου υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται άλλη παρατηρήση που αφορά μικρομεσαίες επιχείρησεις υπέρ κατά απορρίπτεται για ε, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις επίσης υπέρ Κύριε Σιγητά, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις υπέρ κατά ΙΜΚΟ 6652 υπέρ αποχές εγκρίνεται 6650 ήταν τη ΙΜΚΟ 0203-01 τα εργαλεία της ενιαίας αγοράς υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Development of the internal market of goods and services. Un budget 40... Ε, Επιτροπή 4520 τροπολογία 45-20, υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προπολογισμό 45-21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 02-03-04. Ήμκο 66-52. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 02-04-02-03. Γυναικών 64-01. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 04, 03, 01, 05, πράσινη, 54, 51, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 06, 02, 01, 01, τροπολογία τραν και βρασίνων. Ποιοι είναι υπέρ, κατά και ποιοι απέχουν για εγκρίνεται. Τραν, 55, 81 και πρασίνων 470, υπέρ, κατά, αποχες απορριπτωται απορρίπτεται. 06-02-01-02 Πρασίνων 82 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτωται. 08 καινοτομία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 08-02-02-02 γυναικών 64-02 υπέρ κατά Αποχές. Εγκρίνεται. 08, 02, 03, 02, έμβει 54-12 Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. 15-1. 15.02.01 ε, πολιτισμού και βρασίνων. Υπέρ. Ψηφίζουμε αυτό το κονδύλι. Αλλά παρέλειψα ένα άλλο και συμπαθάτε με διορθώνω. Κονδύλι 13.03.12 ΜΕΜΠ 90.02 υπέρ κατά αποχές 15.02.01 όπως είπαμε προηγουμένως πολιτισμού και πρασίνων υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 15.02.01.02 πολιτισμού 61.68 εγκρίνεται πρασίνων 84.56 ενσωμάτωση των ε, προσφύγων εγκρίνεται 33.02.03.01 εταιρικό δίκαιο. Τρεις τροπολογίες. Το ίδιο θέμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Θα ψηφίσουμε τώρα την κατηγορία 1β. Έχουμε μία υπομάδα που είναι πάνω από το σχέδιο προορισμού, έχετε τον πίνακα 2 στο παράρτημα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται η πρώτη ομάδα. Και περνάμε τώρα στις ε, χωριστές ψηφοφορίες. Έχουμε 13 τροπολογίες για την κατάργηση κάποιων κονδυλίων ή για μείωση του ποσού τους σε επίπεδα κάτω 0402 ή 60 ε, και τη 130360 κτλ. Αν δεν έχετε αντίρρηση ψηφίζουμε αυτές τις 13. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτω οι τροπολογίες αυτές. Έχουμε τώρα ψηφοφορίες για διάκριση γραμμών ή για νέε. 21, τροπολογία MEMB 9000 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 130369. Έχουμε δύο τροπολογίες. ECR 8350 badge 4519 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Μετά έχουμε μια σειρά τροπολογιών της ίδιας λογικής. για την ε, ανακατανομή των ε, προσφύγων και για την ένταξη των Ρωμά με αποθεματικα 10-25%. Εδώ ζητώ η κυρία Γκρέσλε να μου πει αν συμφωνεί ότι θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε όλες αυτές τις τροπολογίες μαζί. Συμφωνεί κυρία Γκρέσλε. Ωραία. Σας ευχαριστώ κυρία Γκρέσλε. Ποιοι είναι υπέρ λοιπόν. Διανδάσος χειρός. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Άρα για τα αποθεματικά απορρίπτονται οι τροπολογίες και έχουμε τις παρατηρήσεις. 040260, μια πρώτη τροπολογία μπάτζε 4628 της κυρίας Γκρέσλη. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. badge 4552, Καρθία Θάμπαλ. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 04-0261 μπάτζ 4631 υπέρ. Ναι. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Μπάτζ 4554 54 γκαρδιαθάμπαλ υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 04-0262. Έχουν τροπλία μπάτζ 4630 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 4553 45-53 γκαρδιαθάμπαλ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 040264, τροπολογία της ΓΚΟΥ 7011 και ΜΠΑΤ 4667, Βιέγκας συν συν. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά, αποχές απορρίπτονται. 040601, ΓΚΟΥ 7015, ΜΠΑΤ 4672, υπέρ. Κατά, αποχές απορρίπτονται και σοσιαλδημοκράτη 7707 Poverty Focus. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 13.03.17 για την ολοκλήρωση του European Regional Fund. MEMB 9001. Η συμφωνία της Μάλης Παρασκευής υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 13.03.60. Badge 4601 για τη φιλοξενία των έντονων των Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Μπατ. 4602. Νέα σε τοποθεσία UNESCO. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Και αποχές εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε. Εντάξει, να ελέγξουμε. 13.03. Όχι. Μπάτζ 4602. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται 20 υπέρ, 16, μάλλον 20 κατά, 16 υπέρ. 13.03.61. Μπάτζ 46.03. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Μπάτζ 4604. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Αλλά θα το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρας. Όχι κάποιος. Από το ΕΛΚ. Υπεράριθμος. Να μην ψηφίσει ένας από το ΕΛΚ παρακαλώ. Εντάξει είμαστε τώρα. 37 είμαστε. Εγκρίνεται. 20 υπέρ 16 κατά. 13.62. Έχουμε τροπέ 46 46.05 γκρέσλι. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Μπάτζ 4606 γκρέσλι. Νου UNESCO Sites. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 13.04.60, μπάτζ 46.07. Γκρέσλι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Λοιπόν, πηγαίνουμε Για την κατηγορία 2, ένα πρώτο σου μπλοκ που επαναφέρει τα κονδύλια. Έχουμε το παράρτημα και σχεδόν στον πίνακα 1 είναι τα άγνωτα. ποιοι είναι υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται δεύτερη πομάδα πάνω από το σχέδιο προπολογισμού. Πίνακα 2 του πάρτε του υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται και αυτό το μπλοκ. 0502-0599. Γκουε 7079 τροπολογία υπέρ. μπλοκ θέλετε αλλά δεν γίνεται. Α, το συγκεκριμένο πρέπει να το ψηφίσουμε χωρίς τα υπέρ. Κατά. Αποχές επειδή είναι πάνω από το σχέδιο. Ό,τι είναι κάτω, 05, 02, 09, 08, μέχρι 13, 08, 02, από κοινού, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Στο 34.02.02 έχουμε μια συμβιβαστική τροπολογία υπό ομάδα 2. Ψήφι περ. Κατά. Αποχές. Η γκου 7068 απορρίπτεται, καταπίπτει. Για ξεχωριστές συνέ γραμμές έχουμε το 0504 60 γκου 7075, μπαρ 4673. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Στο 070208 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσωπικών των Ισχυών κτλ. Γκου 7090, Μπατ 4705. Νέα γραμμή αυτή. Νέο κονδύλιο. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 070208, Γκουε 7032, Μπατζ 4704. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Παρατηρήσεις. 05-02-05-99. Έχουμε την ΚΟΕ 70-79 και την ΠΑΤ 46-76. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται. Στη 05-02-08-03 άγκρι, ο 62-12 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Στη 05-02-11-99 μπάτζ 42-43 υπέρ, κατά, δεν είναι σαφές. Θα ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. badge 19 42-43. Ψηφίσατε όλοι. Ένας δεν ψήφισε ακόμα. Πέρασε ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 24 κατά και 11 υπέρ. Να σηκώνετε χέρια παρακαλώ. 05, 03, 01, 01. Single Payment Scheme. Έχουμε τροπολογία FDD 86-05. Υπέρ. Κατά. Αποχές. υπορριπτεται 05, 03, 01, 10. Basic Payment Scheme. FTD 8610 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 05046001 για τη βιώσιμη δραστηριοτική ανάπτυξη. Μπάτζ 4600. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. rubrique 3. Πάμε στην κατηγορία 3. Πρότυπο ομάδα, αποκατάσταση των κοντιλίων σχεδίου. Προπολογισμού πίνακα 1 στο παράρτημα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται δεύτερη ομάδα που είναι πάνω δηλαδή από το σχέδιο προπολογισμού. Στο πίνακα 2 λεπτομέρειες υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. Έχουμε τώρα τις χωριστές ψηφοφορίες. 16.03.02.03 έως 18.07.01. Είτε να μειωθούν τα κονδύλια είτε να καταργηθούν. Μπορούμε να τα ψηφίσουμε μαζί αυτά. Ποιοι είναι υπέρ. Σηκώστε χέρια. Κατά. Σηκώστε χέρια. Αποχές, σηκώστε χέρια. Απορρίπτονται αυτέ οι τροπολογίε. Πάμε στην 23.03.01.01 συμβιβαστική για την υπομάδα 2 του τίτλου του heading 1α, της κατηγοριας Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Καταπίπτει η γκου 7057. Ψηφίζουμε χωριστές γραμμές, συνές γραμμές. 18.02.01.04. Έχουμε τη δημιουργία ενός νέου κονδυλίου S&D 7661 και ΛΥΜΠΕ 6037 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. Έχουμε 18.03.01.01, 02-03-04, τις τροπολογίες ΛΥΜΠΕ 6055, Σοσιαλιστές Δημοκράτες 76-58, ΛΥΜΠΕ 60-56 και Σοσιαλιστές Δημοκράτες 76-59 ψήφι υπέρ όλων αυτών. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 3302 0101 και 3302-0102. Τροπολογία ΦΑΜΑ 6406. Υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παρατηρήσεις. 09-05-01. Κάλτ 61-46. Σωσίδες Δημοκράτης 76-51. Πράσιν 84-58. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 09-05-05. Έχουμε μια προφορική τροπολία του Συγήτου εδώ. Για την τροπολία Badge 46-17. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 15.04.02 Κάλτ 61.50 Σοσιαλιστή δημοκράτη 76.52 Πράσινο 84.57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 16.03.01.03 Μπάτζ 46.19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16.03.01.04 ΑΦΚΟ 67.39 υπέρ κατά αποχές γκρίνεται 16.03.04 κάλτ 61.11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17.04.02 μπάτζ 47.56 γκουε 70.54 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 17 17.04.04. Ένβη, 54-05 Ψήφι Πέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται και κατά πίτη γκου 70-55 και η μπάτς 47-57. Στη 18-02-01-02 έχουμε την μπάτς 42-05 ψήφι πέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 18.02.01.02 μπάτζ 45.23 συγγνώμη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18.04.01 πρώτο που λέει υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Αύκο 67.41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18.04.01.02 αύκο 67.30 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έχουμε την badge 4531 για το κόστος αποζημίωσης. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 33-02-01, γκουε, 70 μπάτζ, 47-66, υπέρ. Κατά, Αποχέ. Απορρίπτονται. Στη, στο κονδύλιο 33-02-02, δύο τροπολογίε. Η πρώτη, άλντε, 77-85, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και δεύτερη είναι 2, η ΦΑΜ 6408 και η πράσινη 8460. Υπέρ. Κατά. εγκρινονται 33020302 εγκρίνονται. 03 πράσινη 84 Υπέρ. Κατά. Αποχές. 330401 04 6653 για την ψηφιακή νέα αγορά υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Badge 4532 γνώση καταναλωτών πιο ανεπτική στόχη. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Nous en venons à la rubrique. Πάμε στην κατηγορία 4. Τρεις, τέσσερις επομάδες έχουμε εδώ. Πρώτη, αποκατάσταση κονδυλίων, βλέπετε τις λεπτομέρειες στον πίνακα 1, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερη υπομάδα που υπερβαίνει το σχέδιο. Παράρτημα πίνακας 2, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τρίτη υπομάδα. Χαμηλότερο από το σχέδιο και αποθεματικά. Στο παράρτημα πίνακα 3. Ψήφι ΠΕΡ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τέταρτη υπομάδα για τους ειδικούς ε, προσώπους. Βλέπετε τα σχετικά στο πίνακα 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Νομίζω ότι για τη 010306 και ως τη 19030106, όλη τη σελίδα 2, μπορούμε να την ψηφίσουμε. Υπάρχει και 1903 βέβαια που δεν χρειάζεται να ψηφιστεί, αλλά αν συμφωνείτε να τα ψηφίσουμε όλα μαζί. Ποιοι είστε κατά αποχές απορρίπτονται επομένως αυτές τις τροπολογίες 19.03.02 στην επόμενη σελίδα έχουμε την ΚΟΕ 72.69 πάνω από το σχέδιο περ κατά αποχές απορρίπτεται και έχουμε την badge 4304 που είναι κάτω υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 20.02.01 έως τη 06 από κοινού να ψηφίσουμε αν συμφωνείτε κατά αν δεν συμφωνείτε αποχές απορρίπτονται. Και πηγαίνουμε στην 21.02.07.05. Γκουε 71.29 που είναι πάνω από το σχέδιο προπολογισμού. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Μετά έχουμε την badge 4441 την badge 4510 και μια σειρά τροπολογιών από κάτω, από το σχέδιο. Θα μπορούσαμε τις ψηφίσουμε μέχρι την 21.07.01. 21.07.01. Μαζί όλα αυτά. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Έχουμε συμβαστική τροπολογία στο 22.02.01.01. Πάνω από το σχέδιο μου κατά 25 εκατομμύρια. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και η γκου 72-71 καταπίπτει. Τώρα νομίζω ότι θα μπορούσαμε 22-02, 03, 02 μέχρι 22, 04, 01, 04. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται. Συμβαστική τροπολογία στο 22.04.04 κατά 16.620.837 ε, ευρώ πάνω από το σχέδιο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρα το 72-72 της ΓΚΟΕ καταπίπτει. Αν το ψηφίσουμε όλες μέχρι το 22 με την 4 με την 3 4 που απορρίπτονται και τώρα 23-02-02 Γκου 70 ε, πάνω από το σχέδιο απορρίπτεται 23-03-02-02 και Γκου 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται χωστή ψηφοφορία για συγκεκριμένα κονδύλια και νέα κονδύλια. 19.02.03 ΑΦΕΤ 52.23 για νέο κονδύλι υπέρ. Κατά και αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζουμε. Σκοτάικλου. Πέρας. Α, απορρίπτεται. 19-17. Παρατηρήσεις. 13-07-01. Μπόγκε. Έχει αποσυρθεί η τροπολογία. Τώρα πάμε στο 19-02-01. Μπέλτερ. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 19.06.01 της ΑΦΕΤ μια τροπολογία του ΕΛΚ και της Επιτροπής ε, Προϋπολογισμών υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21.02.01 συνεργασία με Λατινική Αμερική ΝΤΕΒΕ τροπολογία 5857 αλλαγή τίτλου πρώτον Υπέρ, κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να στοχεύσει εις τους έχοντες περισσότερη χρία. Υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. Η 21.02.02 συνεργασία με την Ασία. Ντεβε, 59.12. Με μια χωριστή ψηφοφορία ετήσι των σοσιαλδημοκρατών. Πρώτο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Όχι, oh, συμπαράτε λέει ο προεδρο Πρώτα πρώτα πρέπει να ψηφίσουμε στο 21.02.02 την αλλαγή του τίτλου. Υπέρ. Και contre. Κατά. Αποχές. Απολύτως. Είκοσι ε, το ίδιο μάλλον, δεύτερο τμήμα υπέρ κατά και αποχές. Το πρώτο τμήμα έχει ε, απορριφθεί. Για το δεύτερο τμήμα τώρα υπέρ κατά αποχές. απορίζεται το δεύτερο τμήμα. 45-26 για το ίδιο κονδύλι της προπολογισμών ε, ανεξιδρυσκεία και πιστεύω πεπιθήσεις των 21, θρησκευτικές. 21.02.03 λέγει του τίτλου πρώτα. Περ, κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε τις ΔΕΒΕ την 58-58 για το κονδύλι 21-02-03. Πέρασε. Απορρίπτεται. 19-17. δυο τροπολογίες των πρασίνων και των προϋπολογισμών. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται πάλι για το ίδιο κονδύλι προστασία των ε, ευάλωτων και αντισημιτισμός. Υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτωται. 21.02.05 Ντεβε. Πρώτα, αλλαγή του τίτλου. Υπέρ. Κατά. Επαλήθευση. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. 2017. Οι δαπάνες θα πρέπει να ε, τηρούν τα του κανονισμού DCI και κρίση της φτώχειας. Υπέρ, κατά. Να φαίνονται τα χέρια σας όπως τα σηκώνετε. Κατά. Επαλήθευση. Ψηφίζουμε. Tout le monde a voté Apparemment και μία Συμπαθάτε με λίγο αλλά μου είπαν ότι για το κονδύλι 210203 όσον αφορά την τροπολογία των προπολογισμών όσον αφορά την ανεξιθρησκεία και τις θρησκευτικές πεπιθήσεις δεν ψηφίσαμε. Εγώ νόμιζα ότι ψηφίσαμε. Αλλά λένε ότι όχι. Εντάξει, ασχετικά δεν έχουμε καθυστερήσει. Οπότε να ψηφίσουμε την τροπολογία αυτή, δηλαδή των προϋπολογισμών υπαριθμών 45-27. Αυτή δεν είναι. Όχι. 45-28 λέει ο πρόεδρος. 45-28 έγινε. Ψηφίσαμε. Bon, 21 επομένως. Πάμε εκεί τώρα. Συμφωνείτε. Ντεβε. Αλλαγή τίτλου πρώτα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ευχαρίστω να κάνουμε παλέψη, αλλά νομίζω ότι είναι το ίδιο αποτέλεσμα και απορρίπτεται. Βελτίωση του συστήματος παιδείας υπέρ, κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 21, 02, 07, 03. Ντέβε και πράσινη σύστημα υγείας, κοινωνική πρόνοια, πρόσβαση στο SRHR. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Παλήθευση. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Α, απορρίπτεται. 14. Σοσιαλδημοκράτε. 75-53, gender equality. Σοσιαλδημοκράτες. Καταπολέμηση της Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Γυναικών για την ισότητα ανδρών και γυναικών υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21.02.07.04 τροπολογίες Ντέβε και Πρασίνων. Καταπίστευμα. Υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος ψηφίζουμε Πέρας. Α, απορρίπτεται. Λίγη 21.02.07.05 Προϋπολογισμών Σοσιαλδημοκρατών και Πρασίνων Τρεις τροπολογίες για τη μείωση της καταπολέμησης τέλο πάντων της φτώχειας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται κατόπιν της ΔΕΒΕ μια τροπολογία 5916 ετήσι των Σοσιαλδημοκρατών θα πρέπει να κάνουμε χωριστή ψηφοφορία. Το πρώτο. Περ κατά αποχές απορρίπτεται το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Α, αποχές απορρίπτεται. 21.02.08.01 Μία τροπολογία γυναικών αύξηση της ε, χρηματοδότησης για SRHR και να αρθεί το κενό που δημιούργησε η κυβέρνηση Τραμπ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Σοσιαλδημοκράτες. Αύξηση χρηματοδότησης για το SRHR. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται προϋπολογισμών 20% για ΜΜΕ και ιδρύματα διπλής εκπαίδευσης υπέρ κατά Υπαλήθευση. ψηφίζουμε πέρας Εγκρίνεται. 22-15. Έχει υποβληθεί αίτημα των Σοσιαλδημοκρατών για χωριστή ψηφοφορία. Το πρώτο τμήμα. Και την τροπολογία εντεύε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Πρώτο τμήμα απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. για, τη, για τα 50 εκατομμύρια προς την Τουρκία, υπέρ. 21.04.01 ήταν αυτή. Υπέρ κατά εγκρίνεται. Έχουν λοιπόν, 15 εκατομμύρια για δράσεις ε, στην Τουρκία. 15. Παρακάτω. Προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημιουργών ελευθεριών και στήριξη δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων. Οι δημοκρατία έχουν ζητήσει δύο ψηφοφορίε όσον αφορά την τροπολογία του προπολογισμού 45-29. Για το πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 22-02-03-02. Αφέτ. 53-51. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται σοσιαλδημοκρατών 75-65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται προγράμματα προγράμματα περισσότερων χωρών περιφερειακή συνεργασία ΑΦΕΤ και ΑΛΔΕ συμφιλίωση στα Δυτικά Βαλκάνια. Υπέρ. Κατά. Α, αποχές. Εγκρίνεται. 22.04.004 προϋπολογισμών όσον αφορά ε, την καταπολέμηση της χρηματοδότησης μίσους ε, τρομοκρατίας και βίας υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 23.02.01 τροπολογίες της ΝΤΕΒΕ των σοσιαλδημοκρατών όσον αφορά την τομιακή και γεωγραφική ισορροπία. Υπέρ κατά εγκρίνεται. Τώρα προχωρούμε για να ψηφίσουμε τα έσοδα και τα ειδικά εργαλεία. Έχουμε κάποια νέα κονδύλια για τα έσοδα. Πρώτα πρώτα, δύο τροπολογίες που έχουν τον ίδιο στόχο. 70-71 και ένα της προπολογισμών 70-73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Δεύτερη Δεύτερη σειρά τροπολογιών. Γκουε και προϋπολογισμών υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτονται αυτές. Για εδώ τα ειδικά εργαλεία. 040401 EGF. Μια τροπολογιών υπέρ, κατά, Απορρίπτονται. Άλλες δύο τροπολογίες τώρα. Της ε, Άλντε και άλλη μία από την Άλντε. Πιστώσεις πάνω το σχέδιο. 40-72 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 4204 έχουμε από τους προϋπολογισμούς 57 για να διαγραφεί το κονδύλι υπερκατά απορρίπτεται δεύτερη σειρά τροπολογιών από το ECR και τροπολογιών για να διαγραφούν τα ποσά υπερκατά αποχές απορρίπτεται 44 αποθεματικό για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης. Υπάρχει μια συμβαστική από τον εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και καταφύπτει η τροπολογία 42-25 των προϋπολογισμών και της ε, Άλντε, της Ρέτζη και των προϋπολογισμών 09 παρατηρήσεις. 13.06.01. Δύο τροπολογίες για τον ίδιο στόχο της ΑΛΔΕ και των προϋπολογισμών. Θύματα τρομοκρατίας. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Νομίζω ότι έχουμε χρόνο για να ψηφίσουμε αυτό τον κατάλογο που αφορά τα πιλωτικά προγράμματα και τις προπαρασκευαστικές δράσεις. Συμφωνείτε? Πρώτα πρώτα. Έχουμε μια ομάδα τροπολογιών με τις λεπτομέρειες εν παραρτήματι και αφορά αυτές τις προσφυγικέ δράσεις. Θα καταπέσουν, λέει, εάν εγκριθεί, ε, όλες εκτός από αυτές που θα ψηφιστούν χωριστά υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται το παράδειγμα. Τώρα έχουμε τις χωριστές ψηφοφορίες. Το είναι ίδιο στόχο όλες, κατάργηση ή των αριθμών των ποσών ή των κονδυλίων τι λέτε να τις ψηφίσουμε μαζί, εισηγητά. Μάλιστα λέει ο εισηγητής. Ωραία, θα τις ψηφίσουμε όλες μαζί. Και τώρα ψηφίζουμε ποιοι είναι υπέρ να σηκώσουν το χέρι. Κατά. Να σηκώσουν το χέρι. Αποχές. Νομίζω ότι καταψηφίζεται. Ναι, οι τροπολόγες αυτές απορρίπτονται. Αυτά για σήμερα. Οι ε, τη τελική ψηφοφορία όσον αφορά τι πληρωμές πρόκειται να σας αποσταλεί απόψε γιατί αφορούσε, αφορά τέλο πάντων αυτά που ψηφίσαμε απόψε για τις υποχρεώσεις και αύριο μπορεί να ακυρωθεί η συνάντησή μας. Εξαρτάται. Αυτά τα οποία πρέπει να ψηφίσουμε άνετα μπορούμε να τα ψηφίσουμε το πρωί. Μπράβο μας, σας ευχαριστώ που τα πήγαμε τόσο καλά, τόσο γρήγορα στις ψηφορίες. Όλα αυτά φίλονται βέβαια στους ε, εισηγητές που τα είχαν προετοιμάσει αλλά και στους συνεργάτες μας, τους συμβούλους να τους χειροκροτήσουμε γιατί τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Κάποιος θέλει το λόγο για τα διάφορα. Όχι. Πέρα συνεδριάσεις. Θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί. Σε 9 η ώρα.